Good morning, ladies and gentlemen. Good... Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν μ' ακούει. What is going on? Doesn't work. Doesn't... Uh, do you hear me? Με ακούτε, συνάδελφοι. Τίποτα δεν ακούτε. Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να σταματήσετε τις ε, συζητήσεις μεταξύ σας για να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Καλώς ήρθατε στην ε, παλιά μας αίθουσα. Έχουμε περάσει μέρες και μέρες σε αυτή την αίθουσα σε προηγούμενες θητείες του Κοινοβουλίου. Έγκριση τη μείσης διάταξης είναι το πρώτο σημείο. Περιλαμβάνεται η μερίσια διάταξη στο φάκελο που έχετε. Αν δεν έχετε σχόλια, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη χωρίς τροποποιήσεις. Κάποιο είπε από την αίθουσα ότι δεν με ακούτε. Μάλλον δεν με ακούτε γιατί δεν κάνετε και ησυχία. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Δεν με ακούτε ακόμη. Okay. Maybe, maybe you should move here. Okay. Not easy. Yeah. Uh, now it's better. Να ακούτε καλύτερα τώρα που άλλαξα θέση. And the technician is necessary. Ας καλέσουμε ένα τεχνικό. I don't hear myself. Hello. Now it's working. Yes. It... Ωραία, φαίνεται ότι τώρα με ακούτε. Αλλά όχι και πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, μερίσια διάταξη. Συμφωνούμε με τη μερίσια διάταξη. Έχετε σχόλια. Ακόμη δεν είμαι σίγουρος ότι με ακούτε με αυτό το μικρόφωνο. Υπάρχουν διαφωνίες για την προτινόμενη ημερήσια διάταξη. Όχι. Οι ανακοινώσει του Προέδρου είναι πολύ απλές. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στην αρχή της απογευματινής μας συνεδρίασης, της 3, θα συζητήσουμε δύο σημαντικά θέματα για 5-10 λεπτάκια για να ενημερωθούμε με το τι έχει γίνει στη διάσκεψη AFET ITRE για τη συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία που μετά από μια συνάντηση που έγινε στις 31 Μαρτίου και η κυρία Πατρίσια Τόγια ήταν μαζί μου, συζητήθηκαν πολλά θέματα και σας θα σας ενημερώσουμε στις 3 η ώρα για αυτή την συνεδρίαση. Επίσης θα ενημερωθείτε και για την πρώτη συνεδρίαση για την ψηφιακή ένωση που έγινε στις 26 Μαρτίου με μεγάλη επιτυχία. Θα ενημερωθείτε λοιπόν και για την ομάδα εργασία αυτή και για τα δύο σημεία 10-15 λεπτά μόνο. Δεν έχουμε το χρόνο τώρα γιατί τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, αν σα ενδιαφέρει συνάδελφοι, κύριε Έλερ παρακαλώ. Μα δεν με ακούει κανένας. Χωρίς μικρόφωνο, τι πρόεδρος να είσαι. But, but not properly. Sorry? But, but it's not working properly. Δεν είμαι σίγουρος ότι δουλεύει σωστά το μικρόφωνο. Εν συνεχίζουμε. Έγκριση των πρακτικών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων συμπεριλαμβάνονται στο φάκελό σα ε, από τις συνεδριάσεις 23-24 Φεβρουαρίου και 9 Μαρτίου του 2015. Έχετε σχόλια για τα πρακτικά? Όχι. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία γιατί θα αρχίσουμε με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Πρώτη ερώτηση, σα αρέσει η Επιτροπή μα, Παρακαλώ, απαντήστε. Άρχεται η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διεξάγεται αυτή τη στιγμή. δεν δούλευε το δικό μου μηχάνημα. Α, τώρα δουλεύει. Εμένα μου αρέσει η Επιτροπή και ψηφίζω θετικά. We can follow now very quickly. Uh, European για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ε, το πρώτο μας θέμα. Η συγκίδια Κάθλιν Βαν Μπρέμπτ, 536 τροπολογίες και πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1 ε, και 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 256 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 258 υπέρ, πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Ας κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 258 πρώτο τμήμα. Έχουμε μία ψήφο παραπάνω από το ΕΛΚ. συνεχίζουμε να έχουμε μια παραπανήσια ψήφο από το ΕΛΚ. Εντάξει τώρα. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Okay. Uh, uh, part, uh, part Για το δεύτερο μέρος τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 265. Πρώτο τμήμα μόνο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Πάλι μία παραπανήσια ψήφο από το ΕΛΚ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2.66. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Ναι, να το ελέγξουμε, δεν είμαστε βέβαιοι. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Vote is Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δίκιο είχατε. 2,67 ψήφι υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 269. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 270 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 271 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική ψηφορία 3 και 35 υπέρ. Κατά. Αποχε... Ε, εγκρίνεται. 2,77 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2,79 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2,93 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2,95 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 2,95. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 304. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 333 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται μάλλον, αλλά θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6, 19 και 30 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τι ωραία. Ε, συγχαρητήρια για τις συμβαστικές τροπολογίες. 4.29 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 430. Τμήμα 1 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 31 και η 428 μαζί. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 435. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 438 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 441 υπέρ. Απορρίπτεται. Όχι ακόμη. Δεν ρωτήσατε το κατά. Επαναλαμβάνεται λοιπόν για την 441. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4.43 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, αλλά το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 444 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 445 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 445. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Θέλετε να τα ελέγξουμε. Όχι. 36. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε την 36, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 39. Συμβιβαστική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, τις αποχές ξεχνάω. Ναι, τις αποχές ζητώ συγγνώμη. Να, να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε. Την 39, συμβιβαστική τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 447 τμήμα 1. Και συμβιβαστική τροπολογία 7. Ο κύριος Έλε θα ήθελα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Γιατί εμείς ψηφίσαμε υπέρ, αλλά άναψαν κόκκινα τα φωτάκια. Τι αποτέλεσμα είχατε στη ψηφοφορία. Στην 39 έγινε αποδεκτή. Πολύ καλό ήταν το αποτέλεσμα, εγκρίθηκε. Όχι, δεν είναι ότι ανησυχούσα, αλλά εμείς ψηφίζαμε υπέρ, αλλά τα φωτάκια έβγαιναν κόκκινα. Θα μπορούσατε να μας πείτε τα αριθμητικά στοιχεία, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Τις αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε που δεν έχουμε τα νούμερα. 30 υπέρ. Σαφώς υπήρχε πλειοψηφία. Λοιπόν, 447 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 443, ε, όχι, 447 ήταν, εγκρίθηκε. Τώρα 37 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 και 38 υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4,73 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Για την 4,73 Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 474 υπέρ, κατά. Πάλι να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 4,75 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4,95 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Την 4,95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συνδεστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνδεσική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 511 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 512 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 514 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 515 υπέρ, κατά, εγκρίνεται νομίζω. Ή να το ελέγξουμε, ας το ελέγξουμε. Για την 515. Closed. Πέρασε τη Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία, συγγνώμη. 516. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 421 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17 συνδροστική υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Όχι, δεν χρειάζεται, απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά. Να την ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Κάποιο λαθάκι. Ας, το ελέγξουμε, δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 102. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 163. Δεύτερο τμήμα μόνο. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Την 163 ελέγχουμε. Το δεύτερο τμήμα της. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα εντάξει. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τι είχα πει πριν. Μπες περιπτώσει. Συγγνώμη για το λαθάκι. 21 συμβαστική υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται πάντως. Συμβαστική 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 συμβαστική υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 23 συμβαστική υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για την 131. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συνδυαστική 27 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συνδεστική 29 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Απορρίζεται. 159 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 105. Δεν ρωτήσατε τις αποχές. Ναι, για την, για την 161 λοιπόν. Ας ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία την 161. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, ξεχνάω να ρωτήσω για τις αποχές, για να πάμε πιο γρήγορα το κάνω. Τροπολογία 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Είχατε δίκιο. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 166. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 169. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 188 και 189. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο τροπολογίε τη σκέψη 33. Πέρα. Απορρίπτονται. λογική σκέψη 25, τροπολογία 190. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 193. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 193. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα 193 εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. 192. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Κάποιες πολιτικές ομάδες ήταν αναποφάσιστες. Γι' αυτό το κοιτάξαμε τώρα, όμως ξεκαθαρίστηκαν όλα. 194 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 194. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 35. Όχι, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 531. 531. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 196. Πέρας. Απορρίπτεται. 197. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2.19. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 220. Υπέρ. Κατά. Φαίνεται πως εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 36. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 37. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 228. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 53 υπέρ, 5 κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους. Μετά από μεγάλες και μακροχρόνιες συζητήσεις, καταφέραμε να ψηφίσουμε. Συγχαρητήρια λοιπόν. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ψηφοφορία για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού Αριθμός 1 κάθετος 2015. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ίδια εισηγήτρια, 24 τροπολογίες, δεν χρειάστηκαν συμβιβαστικές. Ας αρχίσουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 62 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Η δημοκρατία έχει αποτελέσματα. Κυρία Βαμπρέμπτ, θα θέλετε να πείτε κάτι μετά από την τόσο σκληρή δουλειά. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε πολλές ψηφοφορίες μπροστά μας. Καταρχά θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου σε όλα τα μέλη, κυρίως όμως στου κοιόδες εισηγητέ, διότι ήταν μια πολύ καλή δουλειά αυτή που έκαναν σε τόσο λίγο χρόνο και είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι μια παράκληση προ εσά. Ξέρουμε πως αυτό είναι μόνο το πρώτο στάδιο, πολλά στάδια που έπονται και έπειτα, το επόμενο στάδιο είναι προπολογισμό στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και μπάτζε την επόμενη εβδομάδα. Και ξέρουμε πως υπάρχουν αποκλειστικές αρμοδιότητες σχετικά με το ορίζοντα 2020. Και έχουμε μεγάλη πλειοψηφία σε αυτό, χωρίς αμφιβολία. Και υπάρχει και συμφωνία με τις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Οικονομικών Υποθέσεων. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 152, έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και ξέρω πως έχουν αρχίσει συζητήσεις στις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με το αν έχουμε ξεπεράσει την αποκλειστική μας αρμοδιότητα και είμαι σίγουρη πως δεν το έχουμε κάνει αυτό. Και θα ήθελα να πω και σε εσά, κύριε Πρόεδρε, και στου υπόλοιπου σκιώδει ηγητέ για τι άλλε πολιτικέ ομάδε, πω είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουμε εντό των αρμοδιοτήτων μα και να μεταδώσουμε το μήνυμα πω δεν δεχόμαστε αυτόν τον πολύ καλό συμβιβασμό που ψηφίσαμε σήμερα για το άρθρο 5.1.2. Να σας υπενθυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ πολύ για τα σχολιά σας κύριε Βαμπρέμπτη. Η Επιτροπή Ήτρα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για το άρθρο 5.2 για τους στόχους και τους ε, τομείς επενδύσεων. Το άρθρο 18 που αναφέρεται στον ορίζοντα 2020 και το άρθρο 19 στην διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Και κατά κανόνα αυτά εγκρίνονται στις αρμόδιες επιτροπές χωρίς ψηφοφορία. Όμως υπήρξε και μία συμφωνία, συμφωνία κυρίων ανάμεσα ε, για τα νούμερα του τελευταίου προϋπολογισμού και εσείς το γνωρίζετε γιατί σας ενημερώσαμε. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία με την Επιτροπή Μεταφορών, με τον κύριο Κράμερ. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη. Σε γενικές γραμμές όμως, κυρία Βαντρέμπτ, έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας. Αλλά ας προσθέσουμε και αυτό το σημείο ότι έγινε συμφωνία κύριων και είναι εξίσου σημαντική όσο και όλες οι υπόλοιπες συμφωνίες. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για την εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και τώρα περνάμε στο σημείο 7. Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συγητής είναι ο Φίλιπ Τεμπάκερ από την ομάδα Άιντε. Έχουμε 133 τροπολογίες. 183 και γνωμοδοτήσεις και 25 συμβιβαστικές τροπολογίες. Ας αρχίσουμε. Συμβιβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Στην 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και αποχές. θα σας ρωτάω και για τις αποχές. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Και να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ γιατί δεν βλέπω καλά. 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 79. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. 83. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 84. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Λοιπόν, ας ακολουθήσουμε την κανονική διαδικασία. 86, τροπολογία 86 ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές. Σας ευχαριστώ, εγκρίνατε. 87, ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97. Υπέρ. Το πρώτο μέρος της 97. Πρώτο μέρος λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πρώτο μέρος της τροπολογίας 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος της 97. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 105. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 106. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106, 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά θα κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 129. Πέρας. Εγκρίνεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 132. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Και σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. Είναι δύσκολο να δούμε ποιοι συμφωνούν και ποιοι όχι. 133 λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Τη συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147. Υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 147. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 159. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανείς δεν ξέρει. 172 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 173 και 174 μαζί. Να ταυτόσουμε στις τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. 173 και 174 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μεγάλο λάθος. Δεν πειράζει όμως. 175. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 176. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24. Υπέρ. Κατά.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τροπολογία 22. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβατιστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 1 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. για την Ρέγγι 1. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε για αυτό, αλλά δεν βλέπω χέρια. Ρέγγι 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επιτροπή Προϋπολογισμού ή αγγλικό ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος τροπολογία 2 της Επιτροπής Προϋπολογισμού άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Προπολογισμού 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προπολογισμού 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμού 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια συνάδελφε Ντεμπάκερ για την έλξεσή σας. Συγχαρητήρια και σε όλους τους ε, συναδέλφους, σε όλους τους κοιόδης συζητητέ. Περνάμε στο επόμενο, σημείο 8 περιορισμός ε, των εκπομπών ορισμένων ρήπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Ο κύριος Φέντερλε είναι ο εισηγητής. Έχουμε 185 τροπολογίες και έναν αριθμό συμβαστικών τροπολογιών. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Ένα λεπτό. That's um, Τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Τροπολογία 34. Υπέρ. Λοιπόν, η 75 υιοθετήθηκε και τώρα κάνουμε ένα άλμα και πάμε στην τροπολογία 34. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 74 έρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά εποχές έλεγχος για την 38 άρχεται η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται 41 υπέρ κατά εποχές έλεγχος για το 41. Πέρας. Απορρίπτεται. 42 και 43 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 44. Υπέρ κατά αποχές γκρίνεται εντάξει να ελέγξουμε τη 44 ηλεκτρονικά πέρας εγκρίνεται 40 τμήμα 4 υπέρ κατά εποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια, γιατί δεν βλέπω τίποτα. 45 και πάλι. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 46 και 47 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές γκρίνονται. Συμβαστική ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τεροπολογία 50 υπέρ. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 και 31 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Συμβεβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 108 ηλεκτρονικός έλεγχος για την 108 πέρασε απορρίπτεται. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Για τη συμβαστική 4. Περιμένουμε, ήρεμα. Έχουμε έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Είμαστε τόσο γρήγοροι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εποχές έλεγχος για τη συμβαστική 6. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτει. Τροπολογία 123 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, ολόκληρη ομάδα από την 124 μέχρι την 137 τροπολογίες μαζί. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Πέρας. Πάλι ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Εντάξει. Πέρας. Απορρίπτονται. Τροπολογία. 100... Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 131. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. 133 δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πέρασε. Απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές, να ελέγξουμε για την 134. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για τη 15 ελέγχουμε Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται Τώρα, περνάμε σε σωματική ψηφοφορία 135, 136, 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται να ελέγξουμε. Τρεις τροπολογίες μαζί. Αυτό 13-14. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτονται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά ας το ελέγξουμε. 142. αέρας. Απορρίπτεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. γκρίνεται. Κατόν 90 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 190. Πέρας. Απορρίπτεται. 192. Υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. 191. Υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε για την 194. Πέρας. Εγκρίνεται. 195. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε την 195. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 και τροπολογία 18 μαζί, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 2 υπέρ κατά για να ελέγξουμε τροπολογία 2 πέρας εγκρίνεται 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία διορθώνει ο πρόεδρος για το σύνολο της έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 42 υπέρ, 9 κατά 10 αποχές. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την καλή δουλειά. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο. Ο Χωσέ Μπλάνκο είναι ο συντάκτης νομοδότης, εφαρμογή οδηγία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και τη Συμβουλή 22 Μαΐου 2009 για την αρμόνιση ορισμένων τυχών του δικαιώματο του δημιουργού και συγκοινωνικών δικαιωμάτων στην κοινωνία τη πληροφορία. 134 τροπολογίε και 11 συμβιβαστικέ. Να ξεκινήσουμε. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, 21 υπέρ. Κατά. εποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Τροπολογία 8. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ κατά έλεγχος για τη 16 πέρας εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά Εποχές να ελέγξουμε την 44 παρακαλώ ψηφίστε λήξη εγκρίνεται να σηκώνετε τα χέρια παρακαλώ τροπολογία 45 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελαφώς. Για την 80 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται 48 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε τη 49. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε την 63 πέρας Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά Έλεγχος για την 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. εποχέ, απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 97 πέρας κινείται δεκτή 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά χέρι εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά χέρι εγκρίνεται 122 υπέρ κατά χέρι εγκρίνεται 123 υπέρ κατά Αμποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγγνώμη έγινε ένα μικρό λάθος. Τροπολογία 82. Φαινόν δεν την ψηφίσαμε την 82. Στη σελίδα 8. Κάτω από τη συμβαστική 5. Στη σελίδα 8. Να ελέγξουμε για Μάλλον ελέγξαμε την 82 και δεν έχει ψηφιστεί. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. 82. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Συγχαρητήρια. Καλό αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Πάμε στο επόμενο σημείο. Last. Περνάμε τώρα στην τελευταία ψηφοφορία. Προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται εμπορικών απορρίτων κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους. Συντάκτρια η κυρία Μισελ Γιβαζή. ...280 τροπολογίες και συμβιβαστικές τροπολογίες. Και ξεκινάμε με τη συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101, 102 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, Ας το, ε, το ελέγχουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε. Την 11 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, μάλλον εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ελέγχουμε τη 12 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123, 124, 125 μαζί. Υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 123, 124, 125. Πέρασε της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Για 13 ηλεκτρονική ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131-132 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 133-134 μαζί, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 135-136 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 και 155 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 157 και 158 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 150, 160 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε την 179 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία Πέρας στις Απορρίπτεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές. Τα 178 μπορείτε να ψηφίσετε λίγο πιο ξεκάθαρα. Ας ψηφίσουμε τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία για να το ελέγξουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 180. Συμπεριλαμβανομένη τη προφορική τροπολογία των σοσιαλδημοκρατών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρέπει να πάμε πίσω και να ψηφίσουμε και την 23 όμως. Γιατί η 180 δεν αποκλείει την 23, άρα ψηφίζουμε και την 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά, Ας ελέγξουμε την 191 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ή να, το ελέγξουμε για την 11, για τη συμβαστική τροπολογία 11, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 39. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 216 και 217 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε την 220. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 222. Δεν χρειάζεται να τη ψηφίσουμε τη 222. Γιατί απερίφθη η 44. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν τη 222. Το ίδιο ισχύει και για τη 229. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα Επαναλαμβάνω, αφού απερίφθη η 44 δεν ψηφίζουμε ούτε τη 229. Ψηφίζουμε τώρα τη 230. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 231 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 232 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 233 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 234 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 235 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 236 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σύμβαση και τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 251 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές, ας τα ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 267. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 200, ζητώ συγγνώμη, 276 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 277 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 278 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τη 279. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 59. Ωραία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεδραστική τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, α, κα, συγγνώμη, έκανα λάθος για την 81, να ψηφίσουμε πάλι υπέρ, κατά,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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91. 91, ναι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 46 υπέρ, 5 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα σύντομο διαλυματάκι μετά την ψηφοφορία. Εγώ τουλάχιστον χρειάζομαι. Θα ζητήσω από την κυρία Πατρίσια Τόγια, πρώτη αντιπρόεδρο, να έρθει να προεδρεύσει την υπόλοιπη πρωινή συνεδρίαση. Και ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε όχι μόνο τώρα αλλά και στις τρεις. Ευχαριστώ Πατρίτσια. Αν ε, μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας, ε, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, παρακαλώ να το κάνετε γρήγορα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις πρωινές μας εργασίες. Το επόμενο σημείο στην ενημερωσία διάταξη αφορά την γαλαζία οικονομία. Έχει να κάνει εδώ με την εξέταση του σχεδίου έκθεσης που προετοιμασεί ο κύριος Φερέιρα. Καταρχήν θα έδινα το λόγο στον εισηγητή για την έκθεσή του και κατόπιν ε, θα ακούσουμε τους Κιώδης και τους υπολοιπούς συναδέλφους. Ζωάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένες κύριες ιδέες αυτού του σχεδίου έκθεσης πολύ σύντομα. Καταρχήν, Μία πρώτη ιδέα είναι ότι η έννοια της γαλάζιας οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, πολλές οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη θάλασσα και τους ωκεανούς. Συμπεριλαμβάνονται εδώ και παραδοσιακοί τομείς, ή πιο παγιωμένοι τομείς και αναδυόμενοι τομείς. Εδώ αναφέρονται ορισμένοι τομείς ε, οικονομικής δραστηριότητα και στην ε, έκθεση γίνεται και μια αναφορά στο περιορισμένο πεδίο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει σε ένα ευρύτερο και σε μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των προκλήσεων της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας το σύνολο των ποικιλών τομέων που καλύπτουν τη γαλάζια οικονομία. Δηλαδή μια προσέγγιση που να καλύπτει όλες τις τομεακέ και διατομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις θάλασσες, με του ωκεανού και με τις παράκτιες ζώνες. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν συμβαίνει σήμερα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επικεντρώνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων. Μια δεύτερη ιδέα έχει να κάνει με την έλλειψη γνώσης σε σχέση με τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ο περιορισμός ε, αυτός ε, επιβάλλει την καινοτομία και την βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων ε, των θαλασσών και των ωκεανών. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε αυτή την έλλειψη γνώσης, να την καλύψουμε με μεγαλύτερη επένδυση και με σταθερή χρηματοδότηση για τη βελτίωση της γνώσης ε, για το θαλάσσιο περιβάλλον με εγγύηση προβλεψιμότητας μακροπρόθεσμης των επενδύσεων αυτών. Και ε, γίνεται και μια αναφορά σε σχέση με τις περικοπές ε, στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 γίνεται μια κριτική σε αυτές τις περικοπές και ζητείται μια αξιολόγηση αντικτύπου για τις περικοπές αυτές κυρίως στους τομείς που συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία ή σε οριζόντιους ε, τομείς που μπορεί να πλήξουν τη γαλάζια οικονομία. Μία τρίτη ιδέα έχει να κάνει με το εξή, με το, τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους πρέπει να είναι του δημοσίου τομέα. Προτείνονται κάποιες συγκεκριμένοι στόχοι και προθεσμίες που έχουν ως στόχο να αυξηθούν τα δεδομένα που έχουμε είτε για τη στήλη του ύδατος είτε για τους έμβιους πόρους είτε για το θαλάσσιο περιβάλλον. Μία τέταρτη ιδέα έχει να κάνει με την έλλειψη εμπειρογνώμων, ε, σε διάφορους τομείς. Είτε πρόκειται για ερευνητές, είτε για τεχνικούς, είτε για μηχανικούς και άλλους. Αυτή η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών αποτελεί εμπόδιο ανυπέρβλητο για την πλήρη εντοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας. Επομένως, είναι απαραίτητο να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα και να ανατρέψουμε τις τάσεις που έχουμε σήμερα. Έχουμε ουσιαστικά υποτίμηση του κοινωνικού και επαγγελματικού στάτους αυτών των επαγγελματιών και μπορούμε να μιλήσουμε γενικά για αποεπένδυση στους ε, τομείς της εκπαίδευσης και της επιστήμης στα διάφορα κράτη-μέλη. Μια πέμπτη ιδέα είναι ότι ε, το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας ε, δεν θα πρέπει στους ωκεανούς και στις θάλασσες να χρησιμοποιήσει μοντέλα ανάπτυξης που αποδείχθηκαν ανεπαρκή και μη βιώσιμα στην ξηρά. Δηλαδή η έρευνα των πόρων στις θάλασσες και τους ωκεανούς θα πρέπει να σέβεται την κοινωνικότητα να διασφαλίσει μια καλή διαχείριση και διατήρηση των πόρων. Μάλιστα τα ποσοστά της χρήσης ε, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό της φυσικής αναγέννησης ε, των πόρων αυτών. Όταν μιλάμε για πόρους που δεν ανανεώνονται. Επίσης, σημειώνουμε τη σημασία της οικοκοινοτομίας, ε, της κυκλικής οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης των πόρων. Πρόκειται για αρχές που θα πρέπει να εντάσσονται σε όλα τα εφιστάμενα προγράμματα που αφορούν τη γαλάζια οικονομία. Μία έκτη ιδέα είναι η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο κατάλληλο για να παρέχει κίνητρα στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ένα τέτοιο πλαίσιο που να διαρθρώνει υφιστάμενα μέσα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά μιλάμε για την καλύτερη διάρθρωση των υφισταμένων δηλαδή των διευθυντικών ταμείων και των επενδύσεων. Έχουμε και το πρόγραμμα επενδύσεων και να προβλέψουμε καλύτερη προσαρμογή αυτών των μέσων στις αναγκαιότητες που έχουν οι επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς, οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ πέρα από το να υπάρξει, δηλαδή, μιλάμε δηλαδή για την, ε, να εκμεταλλευτούμε τις υφιστάμενες ευκαιρίες. Μία επιπρόσθετη δε έβδομη είναι η αναγκαιότητα στρατηγικής εξειδίκευσης έχοντας κατά νου την ανάδυση και αξιοποίηση των ε, αλυσίδων αξίας, ε, αλυσίδων αξίας που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία. Μία τελευταία ιδέα που θέλω να υπογραμμίσω είναι η σημασία των ε, ε, κοινοτήτων ε, στα νησιά και στις παράκτητες περιοχές. Πρέπει να συμμετέχουν οι κοινότητες αυτές στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις, όλα τα στάδια ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας. Είναι απαραίτητη η προπόθεση για να ελοπιθεί κάθε δυναμικό καινοτομία, δημιουργία θέσεων εργασία, ευημερία και αηφόρου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας. Και για να κλείσω, να προσθέσω το εξή εντός ε, φυσικά των περιορισμών που γνωρίζετε προσπαθεί να γίνει και μια σύντομη τομεακή προσέγγιση. Επικεντρωνόμαστε σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς, διδοκολέργεια, αλία, μεταφορές, εμπορική ναυτιλία, ε, ναυπηγία, διάβρωση των ακτών, ενεργειακή πόρη, ε, έρευνα των ορυκτών πόρων και βιοτεχνολογία. Και γίνονται και κάποιες σύντομες συστάσεις σε σχέση με καθέναν από αυτούς τους τομείς. Η καινοτομία δεν μπορεί και δεν ε, πρέπει να εξυπηρετεί μόνο τους ε, αναδυόμενους ε, τομείς, βιοτεχνολογία παραδείγματος χάρη, έρευνα το θελασσιβητό, αλλά πρέπει να βοηθά και τους παραδοσιακούς τομείς όπως η αλία, η ναυπηγική, η επισκευή των πλοίων. Θα πρέπει λοιπόν να να αναφέρω ότι είχα και μια πολύ καλή επαφή με ε, το συνάδελφο εισηγητή από την Επιτροπή Αλίας ε, που ε, έχει συνεισφέρει στις συστάσεις που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας συγχαίρουμε για αυτή την έκθεση. Είναι πολύ πλούσια σε ιδέες και θα δώσουμε τώρα στην κυρία Σπυράκη το λόγο από το ΕΛΚ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Φερέιρα για την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλε για να ετοιμάσει αυτήν την έκθεση. Κύριε Φερέιρα, σίγουρα όμως πρέπει να περιμένετε πολλές τροπολογίες από τη δική μου πολιτική ομάδα, από το ΕΛΚ και σίγουρα θα συμφωνήσουμε πως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να, εστιάσω στα ακόλουθα σημεία τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είχαν τονιστεί περισσότερο. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω ελληνικά σε αυτό το σημείο γιατί θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στους Έλληνες. Καταρχάς... το report διατύπωσα ότι έχει πέσει σημαντικό βάρος της ανάλυσης σε παραδοσιακούς τομείς που υπάγονται στην λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη στο Blue Growth. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι απαραίτητα κακό. Ωστόσο προβληματίζομαι γιατί συν της άλλης, η προσέγγιση που ακολουθείται είναι προσανατολισμένη στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του status quo σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η έννοια της γαλάζιας ανάπτυξης. Αυτό φαίνεται να γίνεται με μία διάθεση προστατευτισμού Χωρί να υπάρχει κάποια σαφή αναφορά σε τρόπου που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στους τομείς του, της, της γαλάζιας ανάπτυξης ενισχύοντας την οικονομία της αγοράς. Θα σας αναφέρω κάποια παραδείγματα σε ό,τι αφορά τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής. Εδώ γίνεται αναφορά σε παραδοσιακού τομείς της κατασκευής αλλά και της επιδιόρθωσης των πλοίων. Δεν βλέπω κάποια αναφορά στον τομέα της τροποποίησης τους είναι το λεγόμενο retrofitting, είναι ένας τομέας που συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση, στην ανάπτυξη της καινοτομία και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, βλέπω ότι εκφράζεται ένας προβληματισμό για την έρευνα και τους διαθέσιμους πόρους, Παραγωνίζεται όμως το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια σαφή στρατηγική σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων που ενισχύουν τη γαλάζια ανάπτυξη, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου, αγνοείται πλήρω η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ω εργαλείο άντληση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα και από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία θα είναι ακριβώ στοχευμένα στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Το επόμενο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ έχει να κάνει με το στρατηγικό σχεδιασμό των χρηματοδοτικών αναγκών που υπάγονται στο Blue Growth των χρηματοδοτικών τομέων. Κατανοώ την ανάγκη όλοι οι τομεί να πάρουν χρήματα, εύχομαι να γίνεται να παίρνουν όλοι αρκετά λεφτά και μάλιστα άμεσα. Όμως η πραγματικότητα επιτάσσει στοχευμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας και με προσανατολισμό στους τομείς που αναδύονται στην πλέον οικονομία, οι οποίοι δείχνουν να έχουν και τη μεγαλύτερη δυναμική. Θεωρώ δηλαδή ότι θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο λίγοι τομεί και καλύτερο αντίκτυπο να συγκεντρώσουν τον κύριο όγκο τη χρηματοδότηση παρά να πάρουν όλοι από λίγα χρήματα και το αποτέλεσμα να είναι μειωμένο παντού. Κατά τη δική μου γνώμη, οι τομεί αυτοί είναι η βιομηχανία, η ενέργεια, οι εξορίξει, η έρευνα και ο τουρισμό. Και εδώ ακριβώ θα ήθελα να επισημάνω και το τρίτο και τελευταίο σημείο που πιστεύω πω πρέπει να δούμε σε σχέση με το Blue Growth και αυτό δεν είναι άλλο από τον τουρισμό που είναι μοχλό ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία. Ο τουρισμός, όπως δείχνουν τα στοιχεία, δημιουργεί πάνω από 5% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Μιλάμε για 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, για 2,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Ο πολιτιστικός τουρισμός, παραδείγματο χάρη, αντιστοιχεί περίπου στο 40% του πανευρωπαϊκού τουρισμού και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τον αναδείξουμε και στον τομέα του Blue Growth. Το 1 τρίτο όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη προέρχονται από το θαλάσσιο και τον παράκτιο τουρισμό. Και σας λέω μόνο ότι ενδεικτικά πρόκειται για 3,2 εκατομμύρια εργαζομένους που απασχολούνται στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, μια βιομηχανία που συνεισφέρει πάνω από 183 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θα πω κάτι τελευταίο, γυρίζοντας πάλι στα αγγλικά. For all of us... Για όλου εμά ανεξάρτητα από το ποια πολιτική ομάδα προερχόμαστε, μπορεί να συμφωνούμε με τον τρόπο και να διαφωνούμε μάλλον με τον τρόπο, αλλά έχουμε ένα κοινό στόχο. Δημιουργία περισσότερων θέσεων ανάπτυξη και βιώσιμο, ε, απασχόλησης και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να ε, πάνε οι τροπολογίε. Θα ήθελα ξανά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Φερέιρα και ανυπομονώ για μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστούμε. Εγώ δεν έκανα αναφορά στο χρόνο γιατί θεώρησα ότι θα ρυθμίσετε από μόνοι σας. Το χρόνο όμως ε, θα ήθελα να προλάβουμε να κάνουμε και το επόμενο σημείο. Έτσι λοιπόν προσπαθήστε να είστε πιο σύντομοι. Ντάλι για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή κύριο Φερέιρα για αυτό το σχέδιο έκθεση, το οποίο κατά τη γνώμη μου υπογραμμίζει τα κυριότερα ζητήματα. Σήμερα θα ήθελα να εστιάσω σε ορισμένα νευραλγικά σημεία, πέντε τον αριθμό και ορισμένε προτάσει, τι οποίε θα ήθελα να υποβάλω και ελπίζω να τι λάβει υπόψη τη η Επιτροπή. Καταρχά, όταν κάνουμε λόγο για ευρωπαϊκού ωκεανού, ευρωπαϊκέ θάλασσε, να σα πω ότι μιλάμε για κάτι ε, με μεγάλη πολυμορφία. Έχουμε από τον Ατλαντικό, τη Μαύρη Θάλασσα στη ε, Ρουμανία, τις κρύες θάλασσες της Ακτικής και τα ζεστά νερά της Μεσογείου. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαφορές και είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ε, υιοθετήσει μία πολιτική unisex. Επίσης, θα χρειαστεί να γίνει υποδιέρεση των θαλασσών σε ζώνες και κάθε ζώνη θα πρέπει να έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και τις δικές της ε, πρωτοβουλίες και προτάσεις για λύσεις συμφωνώ με τον εισηγητή για το ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάπως ασαφές, όμως πιστεύω πως αυτή είναι η ευκαιρία μας για να έχουμε έναν ισχυρό αντίκτυπο και να δημιουργήσουμε μια στρατηγική που θα μας οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Διότι αυτός είναι ένας ε, τομέας που έχει τεράστιο ανακμετάλλευτο δυναμικό. Η δική μου ομάδα θα υποβάλει τροπολογίες που για παράδειγμα θα συνδέσουν τους ωκεανούς και τις θάλασσες με την ενέργεια. Ιδιαίτερα μια που γίνεται λόγος για ενέργεια και καινοτομία, διότι εκεί υπάρχει μεγάλο δυναμικό το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Ε, τρίτον, ο εισηγητή αναφέρεται στην ανάγκη εντοπισμού χρηματοδότηση για τη γαλάζια οικονομία. Ποιε επενδύσει χρειαζόμαστε, ποια κονδύλια χρειάζονται και συμφωνούμε με αυτό, όμω πιστεύουμε ότι για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ε, τους ε, τομείς αυτούς, πρέπει τα κράτη-μέλη να διεξάγουν τις δικές τους επιστημονικές ε, αναλύσεις και μελέτες και να δουν το, δικές τους, το δικό τους δυναμικό για την γαλάζια ενέργεια έτσι ώστε να υπολογιστούν καταλήλως και να παρουσιαστούν οι οικονομικές ανάγκες. Επίσης να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σπαταληθούν κονδύλια και να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέταρτον, πιστεύω πως ε, πρέπει να ε, εξετάσουμε την ε, δυνατότητα να ανακηρυχθούν ορισμένοι θαλάσσιοι χώροι ως χώροι χώροι διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να δοθεί η δυνατότητα να αναγεννηθούν αυτοί οι χώροι έτσι ώστε να αγγιηθεί η μέλουσα βιωσιμότητα των ε, θαλασσών. Τέλος, θα ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή Ήτρε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή θαλάσσια υπερυπηρεσία. Αυτό προτείνω διότι πιστεύω πω σε μια υπηρεσία η οποία θα αναλάβει την ευθύνη για τον έλεγχο όλων των ε, τομέων που σχετίζονται με τη θάλασσα θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη. Έχουμε πάρα πολλέ υπηρεσίες που ασχολούνται με τον θαλάσσιο χώρο και δεν είναι καλά συντονισμένες μεταξύ τους. Πιστεύω λοιπόν πως ε, είναι καλό να βρεθούν όλες αυτές ε, συγκεντρωμένες έτσι ώστε να συγκεντρωθούν και όλες οι σχετικές ε, πολιτικές. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι άποψη έχουν γι' αυτό. Αυτά προς το παρόν θα χαρώ πολύ για μια επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδης και ελπίζω να οδηγηθούμε σε μια στρατηγική η οποία θα εκμεταλλευτεί πλήρως το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας. Ευχαριστώ τη συνάδελφο. Μαραγκάλ για τους πράσινους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω σπανικά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τη συνεργασία που είχαμε και τη δουλειά που έκανα ο κύριος Φερέιρα. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος, γιατί ακόμα έχουμε δουλειά να κάνουμε και έχουμε και επιχειρήματα να υποστηρίξουμε, όπως είδατε. Το πρώτο συμπέρασμα για την έκθεση αυτή, σχετικά με την ανακοίνωση της Κομισιόν, είναι το εξής. Ε, μέχρι ποιο σημείο ε, αυτό έχει προσθέμενη αξία για την Ευρώπη. Είναι ένα καλό πρωτοβήμα, αν σκεφτούμε την προσθέσαμε στο κοινοβούλιο μας στην έκθεση, αλλά είμαστε ακόμη μακριά και το λέω για το τελευταίο τμήμα της προλαλήσεως σας, της παρέμβασης της προλαλήσεως σας, είμαστε ακόμη πολύ μακριά από να έχουμε μια αυθεντική ευρωπαϊκή πολιτική για τη θάλασσα στο σύνολό της, Κάθε κράτος μέλος υπερασπίζει τα χωρίδατά του, την αλία του, αλλά τώρα η θάλασσα ως αντικείμενο, ως πραγματικότητα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα μάλλον δεν ε, υπήρξε κάτι τέτοιο και φαίνεται αυτό από αυτή την έκθεση. Γιατί εδώ στην ανακοίνωση της ε, Κομισιόν αρχίζει να καθορίζεται μια νέα πολιτική, ένας νέος ρόλος για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτό. Εδώ όμως υπάρχει μια απουσία που δεν μπορούμε να την δεκτούμε και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό αντισταθμίζεται από τις πολιτικές των κρατών μελών αλλά όχι με το σωστό τρόπο γιατί οι εθνικές πολιτικές ούτε μπορούν να αντικαταστήσουν ε, την ευρωπαϊκή παρουσία ούτε μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, ε, γίνεται εδώ μια αναφορά στην ε, έρευνα και στην εξόριση των ορυκτών πόρων με οικονομικούς ε, στόχους και ουσιαστικά μας λείπει μια, ένα πλήρες ε, και αηφόρο όραμα για το θέμα αυτό που να είναι μόνο οικονομικό. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε και για την προστασία του περιβάλλοντος. Και όπως είπε και συνάδελφος το Λαϊκό Κόμμα, πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση, όμως ε, ε, εδώ πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο συνολικοί στην προσέγγιση μας. Επίσης, έχουμε και την έκθεση σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, jobs and growth και εκεί πρέπει να έχουμε ένα όραμα για μία αηφόρο ανάπτυξη, για μία ευφυή ανάπτυξη. Επίσης, ε, αυτό το deep ε, sea mining ε, πλήττεται από την απάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες ε, άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει επιθετικές πολιτικές σε αυτόν τον κλάδο και η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δική της πολιτική αλλά θα πρέπει να έχουμε μια ενεργή στάση ως εταίρος σε σχέση με το deep sea mining. Επίσης, το όλο θέμα της ε, ενημέρωσης. Και με την ανακοίνωση της Κομισιόν, νομίζω ότι θα πρέπει να διευρυνθεί και να αναπτυχθεί προς τη θετική κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, προσβασιμότητα, πρέπει να μιλήσουμε για τη στήλη του ύδατος και νομίζω ότι θα έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μέχρι να συγκεκριμενοποιηθούν τα πράγματα. Επίσης πρέπει να ε, δώσουμε μία ευφυή εξειδίκευση στις πολιτικές των κρατών μελών και πρέπει να έχουμε κατά νου, όπως είπε και ο κύριος Φερέιρα, να συμπεριλάβουμε όλες τις πολιτικές που υπάρχουν σήμερα για τη θάλασσα. Θα πρέπει και τον τουρισμό να τον καλύψουμε ε, με ένα καθολικό τρόπο και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση που γίνεται στην έκθεση, δηλαδή να δώσουμε έμφαση στην κατάρτιση και στη δυνατότητα να ανοίξει ένα κέντρο καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η κατάσταση καινοτομία είναι δύο σημεία κλειδιά. Σας ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω δεν κατά το χρόνο. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διευθυνσή μας. Ο κύριος ε, Ταμπουράνο έχει το λόγο και θα ζητήσω είναι πάρα πολύ σύντομο. Δεν είναι πολύ σύντομος. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Πάκτσας, σήμερα δεν μπορεί να είναι εδώ, επομένως ε, παίρνω το λόγο στο όνομά του. Το μήνυμά του είναι ότι θα υποστηρίξει την προσέγγιση του εισηγητή στο να συμπεριληφθούν περισσότεροι τομείς όπως προτείνει η Κομισιόν, όπως η Δετοκαλλιέργεια και θα υποστηρίξει αύξηση των επενδύσεων αλλά και μια καλύτερη γνώση και μελέτη ε, του θαλάσσιου περιβάλλοντος ε, και φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της εφορία. Σας ευχαριστώ κύριε Ταπουράνου για τη συνεργασία. Κέλλη con davvero alla brevità. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχοντα συντάξει ο ίδιο μία έκθεση για τον τομέα αυτό, με χαρά μου βλέπω πω προχωράμε. Διότι η γαλάζια ανάπτυξη όχι μόνο έχει τεράστιο δυναμικό, όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού και της αιδατοκαλλιέργειας, αλλά ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πτυχές που αφορούν και τη δική μου εκλογική περιφέρεια. Η μία είναι το πρόγραμμα West Wave, ε, στα πλαίσια του οποίου θα μετατρέψουμε σε ηλεκτρική ενέργεια την ενέργεια των κύματων της θάλασσας. Έπειτα, έχουμε μία ομάδα επιστημόνων, ωκεανολόγων που διεξάγουν έρευνες για την χρήση της ενέργειας. Και όπως είπε και ο εισηγητής, ο, τα κονδύλια από τον ορίζοντα 2020 έχουν μειωθεί. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις έτσι ώστε να αναπτύξουμε βιώσιμες λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κουρασπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Κίνγκς. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον εισηγητή για την έκθεσή του, την οποία άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω πως καλύπτει πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία θεωρούμε και εμείς πάρα πολύ σημαντικά. Ωστόσο, θα ήθελα να διευκρινίσω μία παρεξήγηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογή ε, της ανακοίνωσης για την γαλάζια οικονομία. Δεν είχαμε σκοπό να περιοριστούμε μόνο στην ε, εξόριξη στο βυθό της θάλασσας. Θα θέλαμε με τον όρο καινοτομία να καλύψουμε και τους παραδοσιακούς τομείς ε, της ε, θαλάσσιας οικονομίας όπως την ναυπηγική και την αλληλεία αλλά και τους νέους τομείς, την βιοτεχνολογία για παράδειγμα ή την ενέργεια που, μπορεί να, που μπορούμε να έχουμε από τους ωκεανούς. Επίσης, πώς μπορούμε να καθορίσουμε το πεδίο εφαρμογή, το έυρος της ε, γαλάζια οικονομίας και τα κονδύλια που χρειάζονται. Πιστεύω πως αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία εξετάζουμε και θα ήθελα επίσης να εξετάσουμε περισσότερο το ρόλο μιας ξεχωριστής υπηρεσίας που θα ασχολείται με την γαλάζια ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε εξετάσει ακόμα εσωτερικά και φυσικά περιμένουμε την τελική εκδοχή της έκθεσης για να κάνουμε και τα οριστικά μας σχόλια. Ευχαριστώ. Και πάλι θα δώσω το λόγο στον για μισό λεπτό, γιατί μας πήρε ο χρόνος εξαιρετική κυρία Πρόεδρος, ε, δεν μπορώ να πω και πολλά σε αυτό το λίγο χρόνο που μου δίνετε. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο στη ζήτηση, να τους πω ότι σημείωσα δεόντως τις ανησυχίες σας και τις προτάσεις σας και φυσικά νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια σημεία συνένεσης, υπάρχουν βέβαια και κάποια σημεία αποκλήσεων, όμως ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε με όλους τους σκιώδεις στις προτάσεις που θα ανακύψουν και έτσι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση αυτή που ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί είχαμε και πολύ λίγο χρόνο στη θέση μα. Στην ε, προθεσμία κατάθεση προβληγιών, 16 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο που αφορά την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξει τριμερής διαλόγου. Πρέπει να μιλήσουμε για δύο τρίμερε διαλόγου. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στην κυρία Άντελ Καστίγιο, γιατί θα αναφερθεί στον τρίμερη διαλόγο που αφορά την ψηφιακή αγορά. Παρακαλώ. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, είμαστε σε διαδικασία τριμερούς διαλόγου για τη ρύθμιση του κανονισμού για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Αυτό ε, ο κανονισμός που εμείς εγκρίναμε σχεδόν πριν ένα χρόνο στο Κοινοβουλίο 3 Απριλίου του προηγούμενου έτους ε, και Δυστυχώ δεν μπορούσε να αρχίσει ο Δημήτρη διάλογο επειδή παρενέβησαν ε, οι εκλογέ ε, και άλλα γεγονότα, αλλά κυρίω επειδή και το Συμβούλιο καθυστέρησε πάρα πολύ στο να βρει μια κοινή θέση και επομένω ε, να δώσει την εντολή στην Προεδρία, στην εκμεριτροπή Προεδρία, στην Προεδρία τη Λετωνία στην περίπτωση αυτή. Δεν μπόρεσε λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο παρά την καλή δουλειά τη Ιταλική Προεδρία και τελικά ξεκίνησε ο τριμή διάλογο υπόλοιπη τη Λετωνική Προεδρία. Είχαμε λοιπόν το πρώτο τριμερή διάλογο και ήδη μία σειρά τεχνικών συνεδριάσεων, δύο μέχρι τώρα και θα έχουμε και μία τρίτη. Ο επόμενο τριμερής διάλογος θα γίνει στις 21 Απριλίου, την Τρίτη. Μέχρι τώρα Βρισκτή διαπιστώσαμε. Είμαστε στην εξή κατάσταση. Από τη μία, η Προεδρία ανακοίνωσε από την αρχή ότι από τους ε, τρεις κυρίους πυλώνες ε, αυτού του φακέλου, αυτού του κανονισμού, για το φάσμα, το Συμβούλιο είχε αποφασίσει να μην ε, καταρτήσει κάποια κοινή θέση και επομένως να το απορρίψει ως πεδίο διαπραγμάτευσης σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό. Εμεί επιμείναμε ω Κοινοβούλιο στο πόσο σημαντικό είναι ακριβώς το φάσμα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά Τηλεπικοινωνίων. Η Προεδρία συνεχίζει να επιμένει στο θέμα αυτό και επικεντρωθήκαμε, αν και εμείς επιμείναμε όπως σας είπα για το φάσμα, επικεντρωθήκαμε στην περιαγωγή και την ε, ουδετερότητα του διαδικτύου, που ήταν ε, οι άλλοι δύο πυλώνες. Περιαγωγή και Open Internet Neutrality. Ουδετερότητα ανοιχτού δικτύου. Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι σε σχέση με την ΕΚΟ, μία σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των καταναλωτών που σχετίζονται και με το roaming, με τη εργογή και με το ανοιχτό ίντερνετ ζητήθηκε να ληφθούν τουλάχιστον υπόψη σε αυτόν τον κανονισμό, δεδομένου ότι σε σχέση με όλα τα άλλα ζητήματα δικαιω... περί δικαιωμάτων καταναλωτών, που είχαν αποφασιστεί εκείνη τη στιγμή ότι θα πήγαιναν σε μια οδηγία, η Κομισιόν δηλαδή θα έπρεπε να τα συμπεριλάβει στην οδηγία της καθολικής υπηρεσίας σε οποιαδήποτε, όπως και να έχει, κάποιες ε, τέτοιες πτυχές θα συζητούνταν και σε αυτόν τον τριμερή διάλογο. Τώρα, σε σχέση με την περιαγωγή. Η απόσταση με το Συμβούλιο είναι αρκετά σημαντική. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος του Κοινοβουλίου συνεχίζει να είναι ο εξής. Για τα άτομα που είναι σε προσωρινή περιαγωγή να μην υπάρχουν επιπλέον τέλη όταν ε, χρησιμοποιούν ε, είτε την υπηρεσία δεδομένων, είτε τη φωνητική υπηρεσία, είτε τα μηνύματα. Τώρα, στην περίπτωση του Open Internet Neutrality, της ουδετερότητας του διαδικτύου, η Κομισιόν κατόπιν αιτήματος των δύο μερών, καθώς και εδώ υπάρχει μεγάλη απόσταση, θα παρουσιάσει μια σειρά προτάσεων για να προωθήσει τη συμφωνία. Έτσι έχει κατάσταση. Πρόεδρος, ευχαριστώ Πιλάρ. Καλή τύχη για τη συνέχιση αυτού του τριμερούς διαλόγου. Και πιστεύουμε ότι και την επόμενη φορά θα μας κάνεις μια ενημέρωση. Θα δώσω τώρα στο συνάδελφο ε, και που θα μας ε, μιλήσει για το πώς έληξε ευτυχώς ένας πολύ δύσκολος τριμερής διάλογος. Έτσι λοιπόν το συγχαίρουμε εκ των προτέρων. Παρακαλώ κύριε Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο τριμερής διάλογος για τις της ε, χρήσεις γης ολοκληρώθηκε. Η δεύτερη συνεδρίαση ε, του τριμερούς διαλόγου ήταν, ε, ε, ήταν αρχές της Απριλίου και είχε γίνει μια προσφορά για να κλείσει ο Τριμερούς διάλογος νωρίτερα. Είχαμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο και σε αυτό το κρίσιμο σημείο δεχτήκαμε τη θέση του Συμβουλίου για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς Τώρα έχουμε κάτι το μη δεσμευτικό. Συνολικά πριν από την 1η Απριλίου το ε, Συμβούλιο δέχτηκε ε, την αρχική θέση ούτως ώστε να μπορέσει να ληφθεί κάποια απόφαση στη συνεδρίαση του Απριλίου. Η θέση της Επιτροπής Ήτρε σε όλα τα σημαντικά σημεία ήταν ε, αντικείμενο συζητήσεων. Η τελευταία ανάγνωση είχε γίνει μόνο από την ΕΝΒΙ και υπήρχαν διαφορές ήταν ο Βίλιος Τερκουάντρες ε, ε, και ε, δεν υπάρχουν επιστημονικές παράμετροι για να έχουμε έμεση αλλαγή χρήσης γης. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι το ανώτατο κατόφλι για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς είχε προταθεί 5,6% μετά από δύσκολες ε, συζητήσεις με το Συμβούλιο φτάσαμε στο 7%. Και αυτό βάσει των όσων είχαν συζητηθεί και στην προηγούμενη θητεία όπου δεν υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία. Ε, επειδή υπάρχει ε, ε, ε, προαιρετικό 0,5% για τα μελλοντικά σχέδια και εδώ έχουμε ένα από τα σημεία που δεν πέρασαν. Δεν έχουμε χωριστό υποστόχο για την βιοεθανόλη στην, στην απόφαση της και μετά το 2020 θα υπάρχει κάποια προοπτική κατόπιν Προτροπή της Ήτρε αλλά και άλλων και συμφώνησε και ο εισηγητής επ' αυτού, ζητείται από την Επιτροπή να κάνει μία πρόταση μετά, για τα βιοκάψιμα μετά το 2020. Είναι θετικές οι εξελίξεις, μικρά σημεία μείνανε απ' έξω αλλά οι τριμερείς διάλογοι είναι αποτέλεσμα ε, συμβιβαστικών ε, ε, λύσεων. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό και οι συνάδελφοι από την ΕΝΔΙ δέχτηκαν τα δικά μας επιχειρήματα. Αναμένω λοιπόν θετική ψηφοφορία και αυτό συνιστώ για τον Απρίλιο στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν ήταν πολύ, πιο πολύ άριθμη η παρουσία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτοί οι δύο φάκελοι, τα δύο θέματα και πάλι να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λάγκεν ε, για τη λύση που μας επέφερε, που ίσως δεν θα ικανοποιήσει όλους, αλλά όπως και να έχει ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό ζήτημα. Και καλό κουράγιο στην κυρία Πιλάρδη Καστίγιο. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε στις 3.